τα πρακτικά της χθεσινής συζήτηση και τα κείμενα που ευθύθηκαν στη διάστηση των συναδέλφων υπάρχουν αντιρρήσει πρακτικά. Όχι, άρα τα πρακτικά εγκρίνονται. Κυρίε και κύριοι,